Mes chers collègues, bonjour. On va faire ça. Allez, bonjour tout le monde. Καλημέρα σας. Vous avez l'air un peu énervé ce matin. Σας βλέπω λίγο εκνευρισμένους. Ωραία. Όλα θα πάνε καλά. Κύριε Μιζέριε, τι κάνετε. Καλά. Χαίρομαι. Δεν μας φέρατε τον ήλιο. Allez. La communication de la présidente. Ανακοινώσεις της Προέδρου για τις αποφάσεις των συντονιστών. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε πριν από το καλοκαίρι, λέει η Πρόεδρος και διακόπτη, ε, θα βρείτε τις αποφάσεις των συντονιστών της χθεσινής συνεδρίασης. Τα αντίγραφα έχουν διανεμηθεί και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις πριν από τις 12.30 θα ε, πιστοποιηθούν οι αποφάσεις, θα εγκριθούν. Εξάλλου, σε σχέση με ένα σημαντικό σημείο, της Επιτροπής στο πακέτο για την κινητικότητα σας ανακοινώνω ότι πριν από το καλοκαίρι η Ολομέλεια είχε απορρίψει τις τρεις προτάσεις της ε, Επιτροπής για τις κοινωνικές πτυχές της ε, κινητικότητας και έκαναν απομπή σε μας για επανεξέταση. Οι τρεις αυτές ε, προτάσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο για τις διεθνείς μεταφορές, αλλά και για τις συνθήκες εργασίας των οδηγών. Άρα, σχετίζονται με θέματα με ευρύτατα θέματα όπως την απόσπαση των οδηγών, την ανάπαυση, το χρόνο ανάπαυσης των οδηγών, καθώς και την αγορά και το καμποτάζ. Οι τρεις εισηγητές Βιμ Βαντεκάμπ, Ερτούγκ κυρία Κιλόνεν είναι υπεύθυνη για να μελετήσουν την οδό που θα ακολουθήσουμε για αυτά τα τρία θέματα για να τα καταφέρουμε και να περάσουν οι προτάσεις μας. Μετά από συζήτηση με τους εισηγητές είχαμε, ήρθαμε σε επαφές και την κατάλληλη στιγμή θα υποβάλουν το θέμα αυτό, τις αποφάσεις στην Επιτροπή μας. Εντάξει, ωραία. Και τώρα περιμένουμε σε αυτό που περιμένετε όλοι στις ψηφοφορίες. Θα ήθελα να δούμε κατά πόσο υπάρχει, υπάρχει απαρτία. Ωραία, κάνουμε μία επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχετε όλη την κάρτα σας. Κύριε Βιμ Βαντεκάμπ, εσάς περιμένουμε. Με την ησυχία σας. Δεν περιμένουμε το λεωφορείο, αλλά το τρένο σήμερα. Λοιπόν, βάλτε τις κάρτες σας. Allez, on a quatre personnes en plus qui vont voter aujourd'hui. Έχουμε τέσσερις υπεράριθμους. Λοιπόν, υπάρχει απαρτία. Σήμερα θα κρατήσει πολύ ψηφοφορία. Γεζίνα Μάισνερ για τις ε, λιμενικές ε, εγκαταστάσεις για τα απόβλητα. Αρχίζουμε λοιπόν. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Από το ΕΛΚ υπάρχει ένας υπεράριθμος. Ένας υπεράριθμος. Και θυσιάζεται τον κύριο Κούν. Τι να κάνουμε. Λυπάμαι για σας κύριε Κούν. Λοιπόν, πέρας. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέσε νέα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε παλήθευση, εντάξει. Επαληθεύουμε την 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Κύριε Κούν, ψηφίσατε πάλι. Κάποιος άλλος τότε να συμφωνήσετε μεταξύ σας. Ένας πρέπει να αποσύρει την κάρτα του. Ωραία. Για την 5 πέρας και εγκρίνεται. Έμβη 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 10 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Άρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 96. Πέρας. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, θέλετε έλεγχο. Εντάξει. Ελέγχουμε την 99. Πέρας. Εγκρίνεται. Να με εμπιστεύεστε στο εξής. Λοιπόν, 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πες 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δύο παρόμοιε η 6 και η 23. Θέλετε, τι επαλήθευση θέλετε. Πες 13, ωραία, επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Je ferme le vote. Πέρας. Πες 13, εγκρίνεται. Σήμερα δεν με εμπιστεύεστε, βλέπω. Τρίτη φορά με αμφισβητείτε. Λοιπόν, 6 και 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έμβη 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική. Κυρία Μάισνερ. Θα ήθελα να Υπάρχει ένας άλλος ορισμός για το recreational craft, σκάφος αναψυχής, από 2,5 μέτρα ως 24 μέτρα ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόωσης και ένα σκάφος που δεν ασχολείται με το εμπόριο. Αυτός είναι ο ορισμός των σκαφών αναψυχής σύμφωνα με την οδηγία και πιστεύω πως πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Ποιος είναι κατά της προφορικής αυτής Κανένας. Άρα ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία στην προφορική της κυρίας Μάισνερ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η προφορική. Λοιπόν, 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε παλήθευση. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ένας υπεράριθμος πάλι από το ΕΛΚ. Εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται, κύριε Βιμ Βαντεκάμ. Πάλι δεν με εμπιστεύεστε. Να με εμπιστεύεστε. Λοιπόν, 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 115. Πέρας εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές έμβη MV28 υπέρ. Κατά. Θέλετε επαλήθευση της 123. Ψηφίζουμε λοιπόν την 123. Πέρας και απορρίπτεται. Έμβη 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Έμβη 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρεις παρόμοιες 146, 47, 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Έμβη 20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την MV20. Πέρας. Απορρίπτεται. Τι γίνεται κύριε Βαντάλεν. Τι έχετε σήμερα το πρωί. 87 υπέρ. Βιμ Βαντεκάμπ. Κύριε Βιμ Βαντεκάμπ, σας παρακαλώ πολύ Ας μην μιλάτε με τους διπλανούς κατά τις πληρο... ε, ψηφοφορίες 87 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνε. Merci, Ευχαριστώ, κυρία Γκραπίνη. 88 υπέρ. Με συγχωρείτε. MV21. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα περνάμε. Αμπλοκ 91, 112, 145 και 149. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. MV31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32, 31 και 150. Μετά ΕΜΒΗ MV35, 177, 151. Τις ψηφίζουμε unblock υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ωραία. Θα επαληθεύσουμε λοιπόν. Εγώ έχω χρόνο μπροστά μου. Πέρας. Φαίνεται ότι απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέσω 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δύο ταυτόσημες 170-171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Θέλετε παλήθευση. Ωραία. 178 ηλεκτρονική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Να με εμπιστεύεστε, όπως και τις ασφάλειες εξάλλου. Λοιπόν, υπέρ της 179, κατά αποχές εγκρίνεται. MV36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. MV37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. MV38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν μέχρι 197. Ψηφίζουμε unblock υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε γιατί δεν είναι σαφές από την 188 μέχρι την 197. Ταυτόσιμες, εντάξει. Attention! Attention! Λοιπόν, πέρας. Εγκρίνονται. Διακόσια τριάντα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αμαμό 232. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι σοσιαλιστές δεν ψηφίζουν πλέον υπέρ 232 κατά αποχές εγκρίνεται. 29 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμβη 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 233 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο παρόμοιες 234-35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο παρόμοιες 30, 237 πες 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 240 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 200... 241. Θέλετε να υπαλληθεύσουμε. Ωραία. 241. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 242 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. MV42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες, 43, 44, 45 υπέρ, κατά, Α, με συγχωρείτε. Έχουμε ήδη ψηφίσει. Εντάξει. 2.43, με συγχωρείτε. Α, την έχουμε εγκρίνει. 2.45. Αρνοτού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μικέλε, μιλάτε δυνατά. Και δεν με ακούει κιόλα. 2.52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμφυ 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 2.55 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ωραία, θέλετε επαλήθευση της 256. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες Α, που καταπίπτουν. Εμβι MV51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες. 2,57-58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 2,59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κύριε ε, Βιζολιέ, καταψηφίζετε τη δική σας. Σαν τον κύριο Βίμ Βαντεκάμπ. Βλέπω ακολουθείτε την ίδια πορεία. Συνεχίζουμε. 2,60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτε 2,61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο παρόμοιες. 263, 64, 65. Ψηφίζουμε τις τρεις υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Επαληθεύουμε, άρχεται η ψηφοφορία για τις τρεις. Πέρας, εγκρίνονται. 266 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ωραία επαληθεύουμε 267 πέρας απορρίπτεται 268 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πολλές παρόμοιες, MV1, 52, 53, 54 και 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Επαληθεύουμε. Έλεγχος. Πέρας. Και εγκρίνεται. εγκρίνεται. Πες 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρεις παρόμοιες μέχρι την MV55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 271 πέσει 28 MV56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Πες 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρεις παρόμοιες μέχρι την MV2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. MV3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε έλεγχο ελέγχουμε την 32 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές Έμβη NV4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 αποχές απορρίπτεται. Πες 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμβη 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έμβη 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά, αποχές Εμβι MV10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές Εμβι MV8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ άμε συγχωρείτε καταπίπτει 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MV9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MV11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 παρόμοιες 46-47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Ωραία. Κύριε Κράμερ, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνονται. Compromis 8 και πουρ. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμβη 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατά Καταπίπτει 70-71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές Έμβη MV18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμβη 19 Θέλετε να επαληθεύσουμε την 75, ωραία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. MV19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε ε, τελική με ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία για την τελική Allez, je ferme le vote. Πέρασε. 46 υπέρ κατά δύο καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Μάισνερ. Άρα, ε, για να μπούμε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. 46 υπέρ, ένας. Κατά, μπράβο κυρία Μάισνερ, συγχαρητήρια. Μπαίνουμε στη διαδικασία διαπραγμάτευση. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Là. Allez, nous continuons les joies du vote. Oui, monsieur Muselier κύριος Μιζολιέ. Για τη νέα έκθεση. Για ένα θέμα διαδικαστικό. Είμαι σκιώδης για το ΕΛΚ, για αυτή την έκθεση. Εδώ και ένα χρόνο εργαζόμαστε για αυτό το θέμα και μετά τους συμβιβασμούς φαίνεται ότι ότι πέρασαν ε, συμβιβαστικές από τον εισηγητή. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο ή όχι. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι σύνηθες, άρα με εξέπληξε αυτή η οχι εν παση δεν ειναι συνηθες αρα με εξεπληξε αυτη η μεθοδος με τις εναλλακτικές τη στιγμή που είχαν γίνει συμβιβασμοί πριν. Αυτή η διαδικασία με ξένησε κάπως, δηλαδή ότι οι σκιώδεις δεν γνώριζαν τις εναλλακτικές και στη συνέχεια ε, χρειάστηκε να γίνουν συμπληρωματικές. Ευχαριστούμε κύριε Μιζολιέ. Αυτό το είπαμε και χτες. Το είπε ο κύριος Κράμερ η μέθοδος ε, δεν είναι καλή, αλλά ε, θα δούμε τι θα γίνει με τις συμβιβαστικές. Οι άλλοι σκιώδεις δεν το γνώριζαν. Τώρα, ως προς τη διαδικασία έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε εναλλακτικέ συμβιβαστικές οι οποίες θα ε, τεθούν σε ψηφοφορία. Λιντεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ισχύει πω ε, δεν είχαν ενημερωθεί οι σκιώδει ηγητέ. Ενημερωθήκαν. Του στείλαμε τα σχετικά έγγραφα, αλλά θέλω να το πω, να το γνωρίζετε. Η γραμματεία και η διοίκηση βρίσκονται εδώ για να υπηρετούν του ευρωβουλευτέ και όχι να του κατευθύνουν και να του λένε τι θα κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν ίσω θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Μητσοτάκη, λέει πρόεδρο. Κύριε Λιμπεράτσκι, ω πρόεδρο τη Επιτροπή Μεταφορών, δεν δέχομαι τα λόγια σα. Λυπάμαι. Είμαστε πολιτικοί ηθήνοντε και πρέπει να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Είναι πολύ εύκολο να κατηγορούμε την διοίκηση. Από τη στιγμή που κάνουμε λοιπόν πολιτικέ επιλογέ, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Όταν λέτε ότι συνεργαστήκατε με του άλλου εισηγητέ ή συνεισηγητέ, και δεν ενημερωθήκατε. Αυτός είναι λόγος ανησυχίας. Μας το είπε και ο κύριος Κράμερ. Τώρα βέβαια εγώ δεν θέλω να αρχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί δεν ήρθαμε γι' αυτό σήμερα το πρωί. Και ούτω ή άλλω αυτή η συζήτηση δεν μ' αρέσει. Κύριε Κράμερ, έχει 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Ναι, θα ήθελα να πω μόνο πως σε όλες τις συζητήσεις συμμετείχε και η Επιτροπή ΙΜΚΟ και δεν ενημερώθηκε για αυτήν την εναλλακτική συμβαστική πρόταση. Είναι παράδεκτο. Ήταν εδώ από την αρχή, συνεργαστήκαμε και μετά τους απέκλεισαν όπως και του άλλους και εισηγητές. Σε 14 χρόνια που είμαι εδώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Ο κ. Μιζελιέ. Δεν θα ξανοίξουμε την συζήτηση. Να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω εσά Πρόεδρε και τον κύριο Κράμερ. Να σας πω ότι δεν είμαι ψεύτης, αναλαμβάνω τι πολιτικέ μου ευθύνε και ευχαριστώ και την ομάδα του ΕΛΚ που μου ανέθεσε αυτό το τόσο σημαντικό φάκελο. Ευχαριστώ κύριε Μεσελιέ. Ωραία, θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Λοιπόν, συμβαστική 1. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα θέτουμε σε ψηφοφορία την 154 154 ξαναλέει ο Πρόεδρος Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική 2α υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική 2β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε τώρα κατευθείαν στην 190 τροπολογία όχι ένα λεπτό, ένα λεπτό λέει πρόεδρος ένα λεπτό, ένα λεπτό σας περιμένω 190 τροπολογία 190 είστε έτοιμοι όλοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 13 πέρας εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 15 ωραία ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 15 άρχεται η ψηφοφορία για την 15 πέρας της ψηφοφορίας έχετε δίκιο εγκρίνεται εγκρίνεται Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Κυρία Γκραπίνη, θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ωραία, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική 3. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 195 συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, και Κορ. Ωραία. Τροπολογία 17. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ήσασταν κάπως ε, δύσκολοι σήμερα, λέει η Πρόεδρος. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Να μου έχετε εμπιστοσύνη, ξαναλέει η Πρόεδρος. Δύο τροπολογίες. 36 και 97. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήμικο 38 38 την κάναμε, 204 κατέπεσε, 39 και 206 υπέρ. Κατά, αμποχές απορρίπτονται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες. 208-209 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ωραία, 210. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Και έχετε δίκιο, απορρίπτεται η 210. Δύο ταυτόσημες, 19-2-11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται πέρας της πληροφορίας απορρίπτεται μάλιστα Οι σοσιαλιστέ δεν ψήφισαν με τον ίδιο τρόπο, λέει ο Πρόεδρο φαίνεται. Καλά, συνέχεια γίνεται αυτό, λέει. Είναι εθισμένοι. Καταψηφίζουν τις ε, δικές τροπολογίες. Βλέπετε τι γίνεται. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο από το να καταγράψω την ε, ψήφο. Δεν κάνω κρίσεις. Ωραία, συνεχίζουμε, λέει η πρόεδρος. 2.13 και ΙΜΚΟ 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική, όχι λέει η πρόεδρος, ΙΜΚΟ 41. ΙΜΚΟ 41 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες. 233 και 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε κατευθείαν στην συμβαστική 7α. 7α, ποιος είναι υπέρ, κατά, ποχές εγκρίνεται. Πάμε κατευθείαν στην 8α. Συμβαστική 8α. Σελίδα 13. 8α. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφώς το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 8α. 8α ξαναλέει πρόεδρος. Α, και εσείς όμως βλέπω είσαστε διχασμένοι, λέει η πρόεδρος. Πέρα της πληροφορίας. Απορρίπτεται. 8β συμβαστική. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. άποχέ. Εγκρίνεται. Πάμε κατευθείαν στην ΙΜΚΟ 60. Ε, πρέπει να γυρίσουμε κάποιες σελίδουλες εδώ. Σελίδα 18. ΙΜΚΟ 60. ΕΜΚΟ 60 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την ΙΜΚΟ 60 πέρας της ψηφοφορίας ΙΜΚΟ 60 εγκρίνεται Πάμε τώρα κατευθείαν στην ΙΜΚΟ 42. Υπέρ. Όχι, διακόπτη πρόεδρος. Καταπίπτει. Καταπίπτει κύριε Σεντέρ. Είμαστε στην ΙΜΚΟ 42 ξαναλέει πρόεδρος. ΙΜΚΟ 42. Όχι. Υιοθετήθηκαν οι άλλες δύο, οπότε καταπίπτουν. 60 a été adopté. Et... Alors, je 60 εγκρίνεται. Οπότε οι επόμενε δύο καταπίπτουν. Οπότε πάμε στην Ήμκο 42. Ήμκο 42. Ετοιμή. Πάμε. Ήμκο 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΥΜΚΟ 7. Απορρίφθηκε 42, η ΥΜΚΟ 42. Οπότε τώρα κανονικά ΥΜΚΟ 7 λέει πρόεδρο. Κύριε Ερική, αρχίζετε να μα διχάζετε εδώ πέρα. ΥΜΚΟ 7, ΙΜΚΟ 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται η ΜΚΟ 7. Πάμε στην ΜΚΟ 8. ΜΚΟ 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 340 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 9α συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την συμβιβαστική 10α. Συμβαστική 10α, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα κατευθείαν στην 11, συμβαστική 11. Όχι ένα λεπτό, λέει η Πρόεδρος. Όχι ένα λεπτό. Έχουμε άλλες δύο, όμως πριν από την 11. Να συγκεντρωθούμε λίγο. 425 ποιος είναι υπέρ. 425 υπέρ. Κατά. 425. Δύο τροπολογίες πριν συμβαστική 11. Μετά 10α τη συμβαστική κυρία Ριβιταλόν πάμε στη 425. Ψηφίζουμε για 425. 425. Θα κάνουμε μια διόρθωση, λέει ο Πρόεδρος, γιατί κάποιες, ε, κάποιες λίστες ε, ψηφοφορίας δεν είναι ενημερωμένες. Στην συμβαστική μόλις εγκρίναμε έχουμε την 424 την οποία δεν ψηφίζουμε. Οπότε πάμε κατευθείαν στην 425. Εντάξει. Γι' αυτό ακριβώς κάναμε αυτή τη διόρθωση. Γιατί και εσείς στην ΕΛΔΕ έχετε το 425 ως τμήμα του ε, συμβασμού που δεν ισχύει. Οπότε χωριστή ε, ψηφοφορία για 425. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 214 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε ως εκ τούτου κατευθείαν στην 37. 37 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 459 υπέρ. Όχι, συγγνώμη. Καταπίπτει αφού εγκρίναμε την 37. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε κατευθείαν στην συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε κατευθείαν στην 499. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 500 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 501 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 503 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 502 υπέρ, Καταπίπτει, συγγνώμη, λέει πρόεδρος, κάνω λάθος. Τρεις ταυτόσημες. 43, 504, 505 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. 506 καταπίπτει. Συμβαστική 14α υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε κατευθείαν στην συμβαστική 15. Α, ah, για y a une petite erreur sur ma liste. Όχι, συγγνώμη, έχω ένα λάθο εδώ στη λιστα ψηφορία. ψηφορίας. 14β, 14β υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ποιο είπε να ελέγξουμε, ποιος. Balais advisor, qu'est-ce qui vous prend ce matin là ε, Τι πάθατε σήμερα το πρωί, κύριε Βαϊστέρ. Μόνο οι βουλευτέ μπορούν να ζητήσουν έλεγχο, έτσι. Συνεχίζουμε. 15 συμβαστική. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Πάμε κατευθείαν στη συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες. 584 και 101 ΙΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 585. Κατά. Υπέρ. Συγγνώμη. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 586 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 586. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 587 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο ταυτόσημες 588-104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται δύο ταυτόσημες 590-591 που καταπίπτουν καταπίπτουν επίσης καταπίπτουν πάμε κατευθείαν στην 592 592 την 105. Ε, περ κατά αποχές εγκρίνονται. Εμικο 106 περ. κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την ΕΜΚΟ 106. ΕΜΚΟ 106. Πέρα τη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίνεται η ΙΜΚΑ 106. Οπότε, καταπίπτουν. Οι επόμενε πάνε στην 597. 597 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 597. 598 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 599 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες 607 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 601 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 602 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 602. Δύο ταυτόσημες. 603 και 604. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για αυτές τις δύο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτονται όντως. ...605 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται... ...606 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται... ...608 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται... Δύο ταυτόσημες 607 και ΙΜΚΟ 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορία απορρίπτονται. 609 και 109 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 612 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 610 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες. 611 και 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Πολλές ταυτόσημες. 613, 111, 614. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 615 και ΙΜΚΟ 112 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 617 δεν θα την ψηφίσουμε, Κατά καταπίπτει. 616 και ΙΜΚΑ 113 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Δύο ταυτόσημες επίσης, 619 και 618 υπέρ. Κατά, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 619 και την 618. Je ferme le vote. Πέρα τη ηλεκτρονική ψηφοφορία εγκρίνονται. Δύο ταυτόσιμες πάλι, 620 και 114 ΙΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 621 και 115 ΙΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 622. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ όχι καταπίπτει λέει πρόεδρος καταπίπτει καταπίπτει μετά και 623 μπορούμε να την ψηφίσουμε 623 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα ελέγξουμε Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 623. Πέρας της ψηφοφορίας και πράγματι απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες 624 και 116 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 625 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 626 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 627 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 628 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κυρία Γκραπίνη θα ψηφίσουμε την 628 αυτό ζητάτε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 628 πέρα της ψηφοφορίας Α, είχατε δίκιο, απορρίφθηκε. 629 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 630 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δύο ταυτόσημες 631 και 117 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο ταυτόσημες 118 και 632 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται διάφορες ταυτόσημες 633 μέχρι 637 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται θα ελέγξουμε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τις διάφορες αυτές τροπολογίες 633 μέχρι 637 πέρα της ψηφοφορίας έχετε μου εμπιστοσύνη απορρίφθηκαν έτσι δεν είχα πει έτσι δεν είχα πει. Είχα πει ότι εγκρίθηκαν, λέει η πρόεδρος. Πω, πω. Έχω τόση αυτοπεποίθηση που κάνω λάθος, λέει η πρόεδρος. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. μαζί με την ΙΜΚΟ, έτσι, με την ΙΜΚΟ 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατά τη δική σας κυρία Γκραπίνη πάμε στην 62. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 62. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η 62. 18. Συμβαστική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε πάμε κατευθείαν στην 76. 76 του κυρίου Μιζελιέ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε πέρα της ψηφοφορίας και όντως απορρίπτεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Κύριε Κράμερ, θέλετε να ελέγξουμε την 1. Τροπολογία 1. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. πέρα τη ψηφοφορία για την 1 και όντω απορρίπτεται. Κοντά το αποτέλεσμα, αλλά απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Θα ψηφίσουμε την 78. Άρχεται. Allez, on ferme le vote. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται η 78, καταπίπτει η 79, πάμε στην βαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107. Ε, συγγνώμη, 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές για τον 87. Θέτουμε σε ψηφοφορία τον 87. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αμποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 20 θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την ΙΜΚΟ 6. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την ΙΜΚΟ 6. Άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Είχατε δίκιο, είχατε δίκιο, στο συγγνώμη λέει πρόεδρος, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Merci. Allez, nous continuons. Compromis 20. Συνεχίζουμε. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται συμβαστική 21 συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 23 κατευθείαν 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 14 υπέρ κατά αποχές δεν μου φαίνεται ξεκάθαρο το αποτέλεσμα ΙΜΚΟ 14 ψηφίζουμε άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Την ΙΜΚΟ 16. πέρας απορρίπτεται δύο ταυτόσημες 124 και ΙΜΚΟ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε κατευθείαν στην τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136 και η ΙΜΚΟ 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 και ΙΜΚΟ 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 και ΙΜΚΟ 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 καταπίπτει, δεν την ψηφίζουμε 140 και έμικο 24 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 140 και έμικο 24 Πέρα τη εγκρίνεται. Τελική ψήφος για την έκθεση στα δικαιώματα των επιβατών άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 39 υπέρ 2 κατά 0 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Allez, nous continuons. Συνεχίζουμε. Oh, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va Allez, on est reparti, Συνεχίζουμε λοιπόν και βρισκόμαστε στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τα βαρέα οχήματα. Euh, Ξέρω τη χαρά σας για την ψηφοφορία. Έχουμε όμως ε, ακόμα και άλλες. Θα ήθελα λοιπόν να μιλάτε χαμηλόφωνα, αν πρέπει να μιλάτε. Si vous voulez discuter, c'est Οι κουβέντες εκτός αίθουσας. Λοιπόν, περνάμε σε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Αρχίζουμε. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ψηφίζουμε την 88 πέρας υπάρχει ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ Maintenant, c'est correct. Je fermer les Mais, bah oui. Maintenant, c'est Allez, c'est correct maintenant. Madame Virkunen, vous allez voter sur votre rapport quand même. Κυρία Βιρκούνεν, θα ψηφίσετε την έκθεσή σας, φαντάζομαι. Πέρας για την 88, η οποία και απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 91. Πέρα εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια πλειοψηφία, αλλά επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Τρία, Συμβαστική τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Επαληθεύουμε. Συμβαστική τρία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98. Αν θέλετε επαλήθευση, επαληθεύουμε. 97. Έχετε δίκιο. Εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 98. Συμφωνώ, ε, κύριε Τέλιτσκα, μαζί σας. Πέρασε. Πω πω, λέει η Πρόεδρος. Τέλιτσκα, κύριε Τέλιτσκα, τι να πω. Αυτά, αυτά έχει η ζωή. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Συνεχίσουμε. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ήξερα ότι θα ζητήσετε έλεγχο. Ωραία. Ελέγχουμε την 100. Αλλά νομίζω κύριε Τέλιρσκα ότι εγκρίνεται. Πέρας. Είδατε, είδατε πώς τα προαισθάνομαι όλα. Με μία, κατά μία ψήφο υπερψηφίζεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102. Α, καταπίπτει. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Για μία ψήφο. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε τη συμβαστική 5. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται δυο ταυτοσημε ταυτόσιμες, 127-28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε γιατί δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πέρας. Εγκρίνονται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δύο παρόμοιες 132-33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 Ωραία, ελέγχουμε την 134. Πέρας. Απορρίπτεται. Έτσι έχουν τα πράγματα. Pardon. C'est Wim Van de Kamp qui me fait rire. J'ai dit c'est la... Ο Wim Van de Kamp με κάνει και, ε, με κάνει και γελάω. Γιατί εγώ είπα αυτά έχει ζωή και μου απαντά η δική σας ζωή τα έχει αυτά, όχι η δική μου. Και μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ Κύριε Κράμερ, τι θέλετε, να επαληθεύσουμε την 140. Ωραία. Έλεγχος για την 140. Πέρας. Απορρίπτεται κύριε Κράμερ. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, θέλετε έλεγχο. Ωραία. 154 ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες, 8 και 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 8 και 9 ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Α, όχι, πίπτη γιατί είχαμε τη 2 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 17. Πέρας, είχατε δίκιο. Απορρίπτεται. Έτσι έχουν τα πράγματα.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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ωραία. 29. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, επαληθεύουμε την 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ε, για την 36. ισοψηφία βλέπω. Malheureusement, C'est Απορρίπτεται, δυστυχώς. Κύριε Βαντεκάμπ, ενοχλείτε όλους τους συναδέλφους. Σταματήστε. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά, επαληθεύουμε, πέρας, απορρίπτεται. Πενιντάινα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά,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 61 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε καλύτερα την 61 πέρας εγκρίνεται για μία ψήφο συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά η οποία και άρχεται και πέρα της ψηφοφορίας 37 υπέρ 8 κατά 37 υπέρ 8 κατά. Ε, κύριε Βιρκίνεν, εγκρίνεται η έκθεση. Συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες για την διάμεση έκθεση για το ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ 2021-2027 σχέδιο γνωμοδότησης. Αν θέλετε να πιάσετε κουβέντα, λέει η Πρόεδρος, κάτε το έξω.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 Συμβαστική 34 επιπρός κάνει λάθος. Μετά συμβαστική 7. Πάμε στην 34. 34. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά αποχές. Διακόπτη πρόεδρος. Δεν τόλμησα καν να πω τι γίνεται αν εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Κύριε Βαντάλλον, όμως τι φάγατε σήμερα το πρωί και διακόπτεται. φάγα τίποτα παράξενο. Πρόεδρε, να ελέξουμε, μάλλον να ψηφίσουμε. Εμείς θέλαμε να ελέξουμε την 30 και το φώναξα, δεν με ακούσατε. Ωραία. Για την 30 ελέγχουμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 30. Πέρα στις ψηφοφορίες για την 30 και ευρέω εγκρίνεται. 34. Τροπολογία 34. Αφού ο κύριος Βαντάλεν είχε από πριν γνώστο αποτελέσματος. 34 λοιπόν ψηφίζουμε. 34 ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 34. Πέρα της ψηφοφορίας. On remercie Monsieur Muselier de faire passer. Ευχαριστούμε τον κύριο Μισελιέ που πέρασε την τροπολογία αυτή. Μπορείτε να ευχαριστήσετε την κυρία Αργοτάλων και τον Μισελιέ. Allez, moment 35. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέξουμε. ωραία. Je ferme le vote. Πέρα τη ισοψηφία απορρίπτεται. Συμβαστική 8, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική. Όχι, συγγνώμη. 42-43 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά τελική ψήφος άρχεται πέρας της ψηφοφορίας 35 υπέρ 4 ψήφοι κατά Συγχαρητήρια κύριε Ρικέ. Allez, nous continuons sur le vote de l'établissement. Συνεχίζουμε για την θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. a pris du retard là. Oui, mais les trois avis après vont allez vite. parce que... Allez, sur l'Agence européenne du travail, vous êtes prêts Για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία, είσαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Για το σημείο 16, έτσι, τη μεσαία διάταξη. Κύριε Βαντάλεν, θέλετε να ελέξουμε. Ωραία, θα ελέξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 23 σχετικά με θέσπιση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας πέρα της ψηφοφορίας 34 κατά τι να κάνουμε συμβαίνουν και αυτά 24, 24. Σταματήστε να κάνετε θόρυβο. 24. Μέχρι την 286. Όλα αυτά τα ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι, λέει ο Πρόεδρος. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ε, τότε εντάξει, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνονται 90 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 90 πέρας της ψυχοφορίας. απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε κατευθείαν στην 100 της κυρίας Ντελή λέει πρόεδρος υπέρ κατά Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ναι, ναι, κατάλαβα λοιπόν, κατάλαβα, κατάλαβα. Ευχαρίστω. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 του κυρίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε να αλλάξουμε. Ωραία για την 102. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Περάς. Εκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Κύριε Τεντίσκα για την 103 άρχεται περάς και η τελίσκα εγκρίνεται παράξενο συνεχίζουμε συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται περάς για την 109 απορρίπτεται είχατε δίκιο 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέλετε να αλλάξουμε για τα 115 ωραία ψηφίσουμε ηλεκτρονικά περάσει απορρίπτεται Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125. Υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 125 περάς εγκρίνεται 126 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίφθεται. συμβιβαστική 2α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά θα ελέξουμε Allez, je ferme le vote. Απορρίπτεται όντως. Θα περάσουμε τώρα στις επιμέρους τροπολογίες. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130. Καταπίπτει. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 καταπίπτει. Και περνάμε κατευθείαν στην συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, λέει η Πρόεδρος. Θα ελέξουμε 140. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε. Ένα λεπτό page 10. Σελίδα 10 στις 147 και 148 τροπολογίες που είναι ταυτόσιμες. Εντάξει. Όχι, δεν καταπίπτει, λέει πρόεδρο. Στην συμβιβαστική 14 δεν περιλαμβάνονται οι 147-148, οπότε πρέπει να τι ψηφίσουμε χωριστά. Είναι δύο τροπολογίες ταυτόσιμες που θέλω σε ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ μάλλον, λέει ο Πρόεδρος. Στην συμβαστική 14 που μόλις εγκρίναμε δεν περιλαμβάνονται οι 147 και 148. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις δύο ταυτόσιμες τροπολογίες πρέπει να τις ψηφίσουμε. λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο της ξαναθέτω ψηφοφορία. Ξαναρχίζουμε λοιπόν για αυτές τις δύο 147 και 148 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται θέλετε να αλλάξουμε ωραία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για αυτές τις δύο τροπολογίες πέρας ε, εγκρίνονται εγκρίνονται. Περνάμε κατευθείαν στην τροπολογία 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 κατά άποχες απορρίπτεται θέλετε να ελέξουμε κύριε Τελή ωραία θα ελέξουμε λοιπόν άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται υπάρχει και άλλη τελή όμως η δικιά μου λιπρός 153 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επανέρχεστε με την 154 κύριε Ντελή, έτσι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάμε κατευθείαν στην 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε για την 168. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά ίσως να κάνω λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Πέρας και όντως απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 Κυρία Σμιτ, θέλετε να ελέγξουμε ποια τροπολογία. 173. 173, ωραία. Άρχεται λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 173. Πέρας. Έχετε δίκιο, κυρία Σμιτ. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται 173. 174. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 175. Υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 175 πέρας Αγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες, 189-190. Υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τις ταυτόσημες 189 και 190. Je ferme le vote, pardon. Πέρας, εγκρίνονται. Δύο επόμενες καταπίπτουν. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 194-195 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 194-195. Πέρας. εγκρίνονται. Οι δύο επόμενες καταπίπτουν 198 υπέρ κατά αποχές Δεν είμαι βέβαιη, αλλά νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα ελέξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για 198. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 14. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100. Α, γιατί 15. Ελέγχουμε. Ωραία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Ανθρωπολογία 199. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για την 199. Πέρας. Η ισοψηφία απορρίπτεται. 23 με 23. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202 ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες 201 και 16. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνονται. 17 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 203. Κύριε Άλουκα, εσείς θέλετε να ελέγξουμε την 17. Ωραία. Ελέγχουμε τη 17. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται η 17. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 204 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές 204 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 15α υπέρ κατά αποχές θα ελέξουμε. θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για 15α άρχεται η ψηφοφορία 15α και έχετε ένα υπεράριθμο Πέρας. 24-22 εγκρίνεται. Πάμε στην 16, συμβιβαστική 16. Όχι, καταπίπτει λέει η Πρόεδρος, οπότε πάμε στην συμβιβαστική 17, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 227 υπέρ κατά να αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε ωραία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για 227 άρχεται πέρας 30 κατά υπέρ 17 Κάπω μπερδευτήκαμε την ψηφορία με την ανάταση των χεριών, λέει πρόεδρος. Απορρίπτεται 227. 228 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά Άποχες απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 232 παρακαλώ. Πέρας. Για την 232. Ισοψηφία. Έλεξα όπως μου ζητήσατε. Α, ισοψηφία απορρίπτεται. 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 234 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε να αλλάξουμε για την 236 ωραία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 236 άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται με μια ψήφο διαφορά 24-23. 237. 237. Όχι 38 όπως υπέρβος. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 237. Υπέρ. Κατά ηλεκτρονικά, λέει η Πρόεδρος. Πέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά 23-22. Πολύ κοντινό αποτέλεσμα. 230... 240 λέει πρόεδρος, πάμε κατευθείαν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 245 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα ελέξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 245 πέρας Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 246 υπέρ. Κατά. Και εδώ πάλι είναι πολύ κοντά το αποτέλεσμα. θέσμα σε ψηφοφορία τη 246. Πέρας. Εγκρίνεται. 247 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 249 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 251. Πέρας. Εγκρίνεται. 253. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε 253. Πέρας. Εγκρίνεται. Είχατε δίκιο. 255 πέρ Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 255. Πέρας. Εγκρίνεται. 254 κατά πίπτη, 256 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται λέει πρόεδρος αλλά θα ελέγξουμε 256 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα ελέγξουμε 18 άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 18 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 258 υπέρ κατά αποχές θα ελέξουμε δεν είναι σαφές 258 πέρας εγκρίνεται να είναι μια γλωσσική τροποποίηση. 20 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την τροπολογία 20 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Όχι, διορθώνει πρώτος. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 259 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 260-261 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται να ελέγξουμε και για τις δύο αυτές ωραία ξεκινάμε πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίνεται έχετε δίκιο περνάμε Την 272. 272-73 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. ...275 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αλλά θα ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 274 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 277 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 279 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 280 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 284 υπέρ, κατά, αποχές, δεν ξέρουμε. Άρα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 285 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 287. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 287 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Ελέγχουμε. 2.87 πέρας απορρίπτεται 288 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 289 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 290 υπέρ κατά απορρίπτεται 291 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 292 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε πέρας απορρίπτεται 293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε Πέρας. Απορρίπτεται. 295. Με συγχωρείτε, 294 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. 295 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. ...296 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτει. 297 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 298 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 299 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 300 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 300. Πέρας και έχετε δίκιο εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες 303 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Είχατε δίκιο. Οι δύο επόμενες καταπίπτουν 28 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 28. πατέρας Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Θέλετε να επαληθεύσουμε κύριε Ερτούγκ την 27. Άρχεται η ψηφοφορία για την 27. Ε, Πέρας. Απορρίπτεται κύριε Ερτούγκ. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ Ωραία, επαληθεύουμε την 1 του εισηγητή. Πέρας απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36. Υπέρ. άμε με συγχωρείτε, πίπτη. Γιατί εγκρίθηκε 33. 34. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 34. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε λοιπόν την συμβιβαστική 8. Είχατε δίκιο, απορρίπτεται. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά μέχρι τέλους θα είναι πολύ πιο απλό. Αλλά θα κρατήσει περισσότερο. Συνεχίζουμε. Συμβαστική 8α υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Γιατί είναι πολύ κοντινό το αποτέλεσμα. πέρας εγκρίνεται. 49 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Οχές. δεν είναι σαφές άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται η συμβαστική ενέ Θα δούμε κάθε τροπολογία λοιπόν ξεχωριστά. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές, ε, κυρία Μπιλμπάου, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, θα ελέγξουμε. πέρας εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγχουμε. 57. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Έχετε δίκιο, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Αλλά να σηκώνετε τα χέρια. tu rigoles. Πέρας. Με συγχωρείτε κυρία Μπιλμπάου, αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια. Αυτή είναι η δικαιολογία που έχω. Είναι δύσκολο. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε. πέρας εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Επαληθεύουμε την 68. Πέρας. Κατά μία ψήφο υπερψηφίζεται. 69 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε ελέγχουμε λοιπόν Πέρας. Και απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία, επαληθεύουμε την 72 κυρία Γκραπίνη. Πέρας. Απορρίπτεται κυρία Κραπίνη. «73 υπέρ» κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος είπε έλεγχο. Ο κύριος Λοτόφσκι θέλετε επαλήθευση την 11. Ωραία. Ελέγχουμε. Αρχίζουμε την ψηφοφορία για τη συμβαστική 11. Πέρας. Εγκρίνεται κύριε Σλοτοσκι. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίνεται. 79. Α, καταπίπτει και η οκτώ... 80 της κυρίας Μπιλμπάου. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 81 αφού το επιθυμείτε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ναι, εσείς φταίτε, δεν σηκώνετε τα χέρια. 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε κυρία Γκραπίνη. Πέρας. Εγκρίνεται. Είχατε δίκιο κυρία Γκραπίνη. 85 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ε, ελέγχουμε την 85 πέρας εγκρίνεται κατά μία ψήφο 86 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την, 60, την 86, συγγνώμη, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρας, απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά, αποχές, δεν ξέρω. Ε, λυπάμαι γιατί δεν ψηφίζεται όπως πρέπει. Λοιπόν, 87 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά γιατί μόνο έτσι ψηφίζεται φαίνεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά επαληθεύουμε την 88. πέρας. Απορρίπτεται η ισοψηφία. 89. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 89. Ωραία. Πέρας και εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί. Χρειάζεστε λίγο χρόνο. Όχι, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 25 ψήφοι υπέρ 17 κατά. Alors, attendez. Monsieur le rapporteur, vous vouliez prendre la parole. Θέλετε το λόγο, κύριε Σιγητά. Ο κύριος Ντέτζεν έχει το λόγο. Ich wollte... Μόνο να παρατηρήσω κάτι. Ε, θα ήθελα να διαγραφεί το όνομά μου από τον κατάλογο ψηφοφοριών. Par mesure de respect, on essaie d'écouter notre rapport. Προσπαθούμε να ακούσουμε τον εισηγητή. Έχετε και πάλι το λόγο. Να παρατηρήσω λοιπόν κάτι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαγραφεί το όνομά μου από τον κατάλογο της τελικής ψηφοφορίας. και από την έκθεση γενικά. Donc, monsieur Άρα αποσύρετε το όνομά σας από την έκθεση. Ωραία, αυτό θα γίνει. Ναι, αυτό ακριβώς πρότεινα. Ευχαριστούμε κύριε Ντέντζεν. Συνεχίζουμε. Je Συγγνώμη, αλλά έχουμε ακόμα δύο ψηφοφορίες και έχουμε αρχίσει πολύ. Λοιπόν, η κυρία ε, Ρεβονταλόν, μας έχετε προτείνει το δικό σας θέμα για το ΕΤΠΑ και τη συνοχή να αναβληθεί για αργότερα. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε για το ε, διάστημα και το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα. Έκθεση Σαλίνη. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Chez les advisors, s'il vous plaît, je vous demandais de faire... Παρακαλώ οι σύμβουλοι να μην κάνουν τόσο θόρυβο. Τρία, υπέρ. Ψηφίζουμε. Αν θέλετε να ε, μιλήσετε, σας παρακαλώ να βγείτε από την αίθουσα. Τρία, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158 και 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε 181 γραπίνη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 80, 189 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ε, ψηφίζουμε την 197 την επαληθεύουμε 197 πέρας εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε 200, στη 214 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε. Την 214 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 248 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 273 υπέρ. Κατά αποχές αποχές εγκρίνεται. Τη συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 294 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 300 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 301 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 302 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 403 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 404 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 314 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρουμε, επαληθεύουμε. Πέρας εγκρίνεται. 315 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 317 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται υπέρ κατά Μικέλε 318 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 61 υπέρ. Αποχές, 319 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 319 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 322 υπέρ. Αποχές απορρίπτεται 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 324 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 325 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 326 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 328 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 331 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 332 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 333 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 79 καταπίπτει γιατί η 78 εγκρίθηκε. 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 ελέγχουμε. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται πολύ, ναι, πρόεδρος. Πολύ. 83 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ. Όχι, συγγνώμη, λέει η πρόεδρος ένα λεπτό. 25, 25 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ 101 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές αλλά διακόπτη πρόεδρος αποχές δεν φαίνεται είναι οπότε ψηφίζουμε τα 114 ηλεκτρονικά περάς πέρας της πληροφορίας και απορρίπτεται 114 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ Α, όχι, καταπίπτει, με συγχωρείτε, λέει πρόεδρος. 118 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 119. Πέρας. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121. 120 ψηφίσαμε λέει πρόεδρος. Ας μην χάνουμε χρόνο. 120 εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Όχι. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλα. Πάμε γρήγορα. 123. Το πρώτο τμήμα λέει πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψήφος για την έκθεση του κυρίου Σαλίνη άρχεται Πάμε J'ai rattrapé pas mal là. Allez. Je ferme le 35 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Σαλίνη για την έκθεσή σας. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Πάβελ Τελίντσκα. Σχέδιο δράσεις για στρατιωτική κινητικότητα. Συμβαστική 1. Υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές λέει πρόεδρος. Δεν είναι σαφές. Δεν σηκώνεται ψηλά τα χέρια λέει πρόεδρος. 10 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Να ελέξουμε για την 32, πολύ ωραία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ή 35. Ή 35 λέει πρόεδρος. 35. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κύριε Μαρνέσκου. Ακτός μικροφώνου κύριος Μαρνέσκου. Μήπως θα μπορούσαμε να ελέγξουμε για το αν ψήφισαμε την 53 και την 54. Οι 53 και 54 δικές σας κύριε Μαρινέσκου περιλαμβάνονται στην συμβαστική πρόταση 4 η οποία ήδη έχει εγκριθεί, εντάξει. Συμβαστική 5 λοιπόν έχει εγκριθεί. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 να παράθουμε στη 57 κυρία Γκραπέν και να λέξουμε ωραία 57 ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ συγγνώμη. Κυρία Γραπίνη, η 57 εγκρίθηκε. κρίθηκε η, η τροπολογία σας κυρία Γραπίνη. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος για την έκδοση του κ. Τελίνσκα. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. χερί μας, λέει πρόεδρος. Πέρας της πληροφορίας. 28 υπέρ, 7 κατά. 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Τελίσκα. Εγκρίνεται η έκθεσή σας. Μετά την ψηφοφορία που διήρκεσε πολύ, θα διακόψουμε για έξι λεπτά για να ξεκουραστείτε λίγο ή να πιείτε έναν καφέ. Υπότιτλοι Authorwave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

Ξαναρχίζουμε ενώπιον κανενός. Σχεδόν, λέει ο πρόεδρος. si να le euh. λοιπόν, αρχίσουμε με την επόμενη έκθεση. Τη έκθεση που εγώ είμαι ο εισηγητής. Υπάρχουν δύο ε, ε, εμπόδια ε, δημοσιονομικού χαρακτήρα, δηλαδή πρέπει να βρεθούν, να εξευρεθούν πιστώσεις και υπάρχει και το θέμα της ε, ρύθμισης από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα και ε, την ρύθμιση περνάνε 8 χρόνια από το ένα στάδιο στο άλλο και πολλά σχέδια έχουν εγκαταλειφθεί γιατί ακριβώς μεσολαβεί ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν λοιπόν για την απλούστευση και την συντόμευση των, ε, της περίοδου που μεσολαβεί για την ελοποίηση του ευρωπαϊκού, διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Έχουν υποβληθεί συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία ενιαία αρχή, μία ενιαία θηρίδα για να βελτιώσουμε η δυνατότητα υλοποίησης και αυτό αφορά και τη διαδικασία διοδότησης και πιστοποίησης και από την άλλη πλευρά η πρόταση της Επιτροπής έχει σκοπό να συντομεύσει στα τρία χρόνια τις ε, διαδικασίες, τις διοικητικές διαδικασίες ε, βεβαίως με το σωστό νομικό υπόβαθρο. Γι' αυτό υποστηρίζω αυτές τις προτάσεις και θα ήθελα να προσθέσω ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα κατεξιοδότηση πράξης προς μία άλλη αρχή έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτή την ενιαία θηρίδα και έτσι ώστε οι περιφερειακές αρχές ή αυτόνομες αρχές να έχουν μία ενιαία θηρίδα. Επίσης υποστηρίζουμε και το ενιαίο δικαίωμα εφαρμογής για τις ε, διασυνοριακές ε, συναλλαγές και μεταφορές, έτσι ώστε να απλουστευτούν οι κανόνες της αγοράς και αναγνωρίζουμε το ότι τα σχέδια που θα ληφθούν υπόψη από αυτή την ενιαία αρχή θα έχουν προτεραιότητα σε σχέση με την ε, έκκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έτσι θα ενισχυθούν και οι προτάσεις της Κομισιόν και φυσικά γνωρίζω ότι θίξατε ορισμένα ζητήματα σε σχέση με την επικουρικότητα. Εδώ υπάρχει πολύ σημαντικό διακύβευμα και αυτός ο κανονισμός είναι πολύ σημαντικός για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα των ε, διευρωπαϊκών ε, δικτύων μεταφορών. Αυτά κύριε, κυρία Πρόεδρε επί του θέματος και να μείνω στα σχόλια των ε, συναδέλφων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βιμ Βαντεγκάμπ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ντομινίκ Ρικέ για το σχέδιο έκθεσης. Σήμερα το πρωί έλαβαν χώρα πολύ σημαντικές ψηφοφορίες και η πρόταση αυτή από την Κομισιόν δεν έχει λάβει την προσοχή που θα έπρεπε. Μάλιστα ακούσαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τα 247 δισεκατομμύρια από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Αυτό οφείλεται σε αρκετές ε, διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν και όμως κάθε φορά που συζητάμε για το δίκτυο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών αναφέρουμε και τις ιδιαιτερότητες του και αυτά που πρέπει να γίνουν, τη γραφειοκρατία που είναι υπερβολική και περιττή, η οποία καθυστερεί την υλοποίηση των προγραμμάτων. Θεωρώ πως θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η μονοαπευθυντική θηρίδα και αυτό πρέπει να επισπευστεί. Πρέπει οι κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση. Η εξοικονόμηση 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναφέρει ο εισηγητής και Κομισιόν είναι μεγάλο ποσό. Και η μονοπευθυντική αυτή η θηρίδα φυσικά θα ε, διαχειρίζεται, θα είναι αρμοδιότητα των ε, εθνικών αρχών, θα υπάρχουν μικρότερες προθεσμίες για τα διάφορα έργα. Θα υπάρχουν έργα με υψηλή προτεραιότητα λόγω του τοπικού τους ε, ενδιαφέροντος και της τοπικής τους σημασίας. Σε γενικές γραμμές λοιπόν συμφωνούμε με την πρόταση της Επιτροπής και με την έκθεση του κυρίου Ρικέ. Ίσως ε, καταθέσουμε ορισμένες τροπολογίες, δεν θα είναι όμως πολλές. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ρικέ για την εισήγησή του και για τα στοιχεία στα οποία επικεντρώθηκε ώστε να, όπως ξέρει και ο ίδιος, να διευκολύνουμε αυτό το εργαλείο το συνδέοντα στην Ευρώπη για να είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Και Όντως υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη για νέους μηχανισμούς. Εγώ πάντως υπέβαλα με τη βοήθεια της Επιτροπής επειδή συνεργαστήκαμε μια ιδέα ώστε ακριβώς να διαμορφώσουμε ένα μηχανισμό που θα κάνει όσο πιο αποτελεσματική γίνεται την αντιμετώπιση αυτών των διασυνοριακών προβλημάτων ώστε να έχουν όλα αυτά υποχρεωτικό χαρακτήρα και σε ένα κοινοτικό πλαίσιο να ξεπεράσουμε τα εμπόδια των ημερών κρατικών σχέσεων. Η αλήθεια δεν μπορούμε να πάμε πέραν της συνθήκης, αλλά όπως λέγαμε, αν δεν μπορούμε να πάμε πέρα από αυτό που λέει η συνθήκη, θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Και να αναζητήσουμε συνταγές αξιολόγησης των προγραμμάτων που συμφώνησαν οι χώρες μέλη στις Βρυξέλλες ώστε να πιέσουμε ακριβώς τις χώρες μέλη που είτε υπερ-υποβάλλουν ή υπο-υποβάλλουν προγράμματα Παρεποδίζοντα την εξέλιξη διασυνοριακών προγραμμάτων που διάφορα από εμάς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για άλλη μια φορά και θα καταθέσουμε αντίστοιχες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σεντέρ, ο κύριος Ζωτοσκή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρικέ για την έκθεση. Η ομάδα μας στηρίζει τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επισπεύσει τις ε, διαδικασίες για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μία ραχοκοκαλιά μεταφορών και η υπερβολική γραφειοκρατία φαίνεται πως είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτό. Πέρα από την έλλειψη πόρων και των ε, διαφορών εμποδίων που οδηγούν στην ε, εκπρόθεσμη ολοκλήρωση έργων. Διασυνοριακά, επίσης, πρέπει να δούμε τις ελλείψεις σε διασυνοριακά έργα. Η υλοποίηση λοιπόν των έργων και η διάδρομη είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό και τα άρθρα 7 και 8 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικά θεωρούμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία και τις ε, διοικητικές διαδικασίες για έργα εντός ενός μόνο κράτους μέλους, έχουμε τις αμφιβολίες μας. Δεν ξέρουμε αν η πρόταση της Κομισιόν θα είναι το ίδιο αποτελεσματική σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν εθνικές διαδικασίες για την έκδοση αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο για μεγάλα έργα υποδομών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως στερούνται λογικής. Για παράδειγμα, Μεγάλη πρόκληση είναι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και λόγω αυτών μπορεί να καθυστερήσει η ολοκλήρωση ενός έργου. Γι' αυτό λοιπόν ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει την ελευθερία να εφαρμόσει τον καλονισμό με τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία του και τις εφιστάμενες δομές του. Θέλουμε δηλαδή να καταργηθούν τα περιτά στοιχεία της διαδικασίας, αλλά να μην καταλήξουμε και στο χάος αυτό θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις και δεν θα επισπεύσει τη διαδικασία. Θα υποβάλουμε και εμείς τροπολογίες και θα ε, συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους. Ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο. Οι διερμηνείς διακόπτουν διότι έχει λήξει το ωράριό του το πρωινό. Η συνεδρίαση συνεχίζεται χωρίς διερμηνία. Also natürlich